ενός συντονισμού με τους διεθνείς εταίρους ώστε να καταλήξουμε σε σταθεροποίηση της χώρας και σε υποστήριξη της πολιτικής διαδικασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Επίτροπο Ρέντινγκ. Ολοκληρώνεται η συζήτηση για το ψήφισμα αυτό. Έξι προτάσεις ψηφίσματος έχουν κατατεθεί και η ψηφοφορία θα γίνει μετά την συζήτηση των ψηφισμάτων. Το επόμενο σημείο είναι το ψήφισμα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Μπαχρέιν και δίνουμε το λόγο στους συντάκτες, ο συνάδελφος Ρέπο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Μπαχρέιν έχει πάρει μια δυστυχή στροφή, μια τυχή στροφή τελευταία ή έχουν κατασταλεί άνθρωποι που διαδηλώναν υπέρ της δημοκρατίας ε, και λαμβάνουμε και ανησυχητικές αναφορές για το τι γίνεται στις φυλακές. Υπάρχει και κριτική ε, που γίνεται στην κυβέρνηση πέρα από τους δρόμους αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Αραβική Άνοιξη έχει υπάρξει ένα κύμα υπέρ της δημοκρατίας ε, στο Μπαχρέιν και εδώ πρέπει να αποφύγουμε ε, την υποκρισία, πρέπει να αποφύγουμε τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, πρέπει να λειτουργήσουμε σύμφωνα με τις αξίες μας, mm. θα πρέπει να ακούσουμε όλα τα τμήματα του λαού και πρέπει να το υπενθυμίσουμε στο Μπαχρέιν αυτό. Εδώ δεν υποκινούμε κάποια επανάσταση. Η πολιτική βία και οι πολιτικοί κρατούμενοι μας δείχνουν ότι στο Μπαχρέιν δεν πάνε τα πράγματα όπως θα έπρεπε. Ο κύριος Τάνοκ. Ο κύριος Τάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτά που έγιναν το 11 στο Βαχρέιν ήταν σοβαρά γιατί η αστυνομία αντέδρασε δυσανάλογα και σκότωσε πολλούς διαδηλωτές. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τέτοια κλίματα πρέπει να δικαστούν. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι από το προηγούμενο κατεπήγον ψήφισμά μας του Ιανουαρίου έγιναν τόσα πολλά ώστε δικαιολογείται και δεύτερο. Πρέπει λοιπόν το κοινοβούλιο μας να είναι άμεμπτο γιατί δεν μπορεί να κατηγορεί τον Μπαχρέιν ενώ αγνοεί ότι υπάρχουν γειτονικέ χώρε που κάνουν χειρότερα πράγματα. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει προχωρήσει προ περισσότερη δημοκρατία από την Αραβική Άνοιξη. Το Μπαχρέιν πρέπει να το συγχαρούμε για την πρόοδο που έκανε ο διάλογος του βασιλέως και πάνω απ' όλα για τον καθορισμό τον περασμένο Ιούλιο ενό διαμεσολαβητή με την αστυνομία. Φυσικά πρέπει να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι για να μπορέσουν όλοι να ασκήσουν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα όπως την ελευθεροτυπία και την ελευθερία του λόγου. Αλλά το Μπαχρέιν τα γνωρίζει αυτά και δείχνει και ενθαρρυντικά στοιχεία προόδου. Ο, η ίδρυση του δικαστηρίου, του Αραβικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν είναι ακριβώς μια τέτοια ένδειξη. Και αυτό ενθαρρύνω όλους τους συναδέλφους να συνάψουν ε, επικοδομητικές σχέσεις με τη χώρα αυτή και διάλογο και όχι να κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας υποκριτικά και να μην βοηθάμε έτσι κανέναν. Ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ. Για δύο λεπτά η κυρία Βεργιά. Όταν διαβάζει κανείς το ψήφισμα βλέπει ότι είναι μετριοπαθές η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Μπαχρέιν είναι ανησυχητική. Οι μεταρρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται και πολύ γρήγορα. Από τον περασμένο Αύγουστο η κατάσταση έχει χειροτερέψει, η καταπίεση χειροτερεύει και οι μεταρρυθμίσεις είναι αντίθετες από αυτές που υποσχέθηκε το κλάν του Χαλίφα. Έχει σκληρινθεί ακόμη περισσότερο η νομοθετική του πανοπλία. Έχουν κατεβεί διαδηλωτές στο δρόμο που ζητούν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και παρόλα αυτά η αστυνομία τους καταπιέζει βία με την απειλή της παρέμβασης του Ιράν. Αλλά όσοι γνωρίζουν την περιοχή γνωρίζουν ότι αυτά είναι μύθοι του καθεστώτος που εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Σουνιτικής δυναστείας εκεί με σύμμαχο τη Σαουδική Αραβία και στις Ηνωμένε Πολιτείε που κυκλοφορούν εκεί τον πέμπτο στόλο. Ο Χαλίφα Μπιν Σαλμάν Αλ Χαλίφα είναι στην εξουσία εδώ και πάνω από 60 χρόνια και τα ελέγχει όλα. Δεν χρειάζονται πια καθυστερήσεις. Επειδή η περιοχή αυτή έχει μεγάλα στρατηγικά συμφέροντα, η διεθνής κοινότητα έχει μεγάλες ευθύνες και πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μπαχρέινη επιδεικνύουν μεγάλο θάρρος. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε ξεχασμένους της Αραβικής Άνοιξης. Δυστυχώς η Ένωση δεν έρεται στο ύψος των αρχών της σε αυτή την περιοχή. Ασχολείται μόνο με συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Δεν μπορεί να αφήσει τους Μπαχρίνι να συνεχίσουν να αλληλοσφάζονται. Γιατί όλοι συμφωνούν ότι είναι κατά του καθεστώτος. Δεν μπορούμε πια να σοπάσουμε. Δεν θα κρυφθούμε αυτό το ψήφισμα γιατί δεν ανταποκρίνεται στις αξίες μας. Και να εκφράσουμε έτσι την αλληλεγγύη μας με το λαό του Μπαχρέιν. Ευχαριστούμε κυρία Βερζιά. Τώρα ο κύριος Λίσεκ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το Μπαχρέι ε, είναι μικρό, αλλά είναι μια πολύ σημαντική χώρα στην περιοχή. Πρόκειται για ένα κράτος ε, είναι, που είναι σαφές ότι δεν είναι 100% δημοκρατικό, αλλά ας ε, λάβουμε υπόψη ότι έχει κάνει κάποια βήματα για την υλοποίηση του δικαστικού συστήματος και της βελτίωσης του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και γι' αυτό θα πρέπει τουλάχιστον αυτό να το λάβουμε υπόψη. Πρόκειται για μια χώρα με την οποία συνεργαζόμαστε και καθώς αυτή η χώρα συνεργάζεται μαζί μας ε, θα πρέπει όχι μόνο να καταδικάζουμε αλλά να αναγνωρίζουμε και τις πρόοδους αυτές ε, και αναφέρονται στο ψήφισμα τα βασανιστήρια που έχουν γίνει στο Μπαχρέιν. Αυτό το καταδικάζουμε. Αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες ε, για το ότι εργάστηκαν επικοδομητικά για την υλοποίηση αυτού του ψηφίσματος. Εμείς νομίζουμε ότι είναι ισορροπημένο το κείμενο και θα χρησιμεύσει για τη μεταρρυθμίση του Μπαχρέιν. Ελπίζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λίσεκ και τώρα η συνάδελφο Χάρκιν μισή λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το ψήφισμα αυτό μεταξύ άλλων τονίζει την κατάσταση στο Μπαχρέιν όπου οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν ε, προσαγωγές, κρατήσεις ε, και ε, ε, καταδίωξη. Ε, λαμβάνουμε υπόψη μας ε, τους γιατρούς, τους δικηγόρους, τους υπερευθυνσίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλους αυτούς που προστατεύουν την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα ήθελα να αναφέρω δύο κρατουμένους, τον Αμπίλ Ρεζά, τον οποίο συνάντησα, και τον Αμπτούλ Χαντί Αλκβάτζι, του οποίου συνάντησα την οικογένεια όταν ήμουν στο Μπαχρένι, ότι εκείνο ήταν φυλακισμένο εκείνη την εποχή. Ο κύριο Τάνοκ ρώτησε αν όντω χρειαζόμαστε ένα ψήφισμα για τον Μπαχρέν. Εγώ θέλω ε, να ε, ε, αναφέρω το θέμα της χρήσης αερίων στο Μπαχρέιν. Φαίνεται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τοξικά χημικά και έχουν θανατωθεί 50 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείται ένα τέτοιο χημικό όπλο θα πρέπει να καταδικάζεται σύμφωνα με τις διεθνείς διατάξεις. Είναι ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο τώρα που γίνονται οι αντίστοιχες συζητήσει για τη Συρία, αλλά φαίνεται ότι έχει αγνοηθεί. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να γίνει άμεσα μια έρευνα στο Μπαχρέιν για τα χημικά ε, όπλα, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα για τη χρήση χημικών όπλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Χάρκιν. Τώρα ακολουθούν οι ομιλητές ε, εκ μέρους των πολιτικών ομάδων, συνάδελφος Πόσελτ. Κύριε Πρόεδρε, το βασίλειο του Μπαχρέιν βρίσκεται ε, στο σημείο που είναι επίκεντρο ε, των βλέψεων ε, του αραβικού κόσμου. Η διένεξη μεταξύ Σουνιτών και Σιητών, οι βλέψεις του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας, οι διενέξεις μεταξύ εθνικιστών και όλα τα γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά συμφέροντα οδηγούν σε μεγάλη ανησυχία για τη σταθερότητα. Θα πρέπει η σταθερότητα να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Χαιρετίζουμε το ότι υπάρχει ένας υπουργό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι υπάρχει ένας διαμεσολαβητής και ότι υπάρχουν προσπάθειες για καλύτερη πολιτική για τις γυναίκες, αλλά θα έπρεπε ο βασιλιάς Ισαλ Γαλιφά να λάβει πιο σημαντικά μέτρα και γι' αυτό αυτό το ψήφισμα είναι δετιολογημένο ε, είναι ε, μετριοπαθές, αναγνωρίζει τις μεταρρυθμίσεις, αλλά ζητά και περισσότερες πρόοδους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πόσελτ. Η συνάδελφος Γκέρινγκ Ντόντενμπεργκ. Ευχαριστώ. Και πάλι βρισκόμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητάμε την κατάσταση στο Μπαχρέιν. Από ό,τι φαίνεται οι αρχές δεν ε, υποχωρούν ενώπιον των πολιτών οι οποίοι ζητούν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Είδαμε ε, ότι είχαμε βασανιστήρια, αιματηρές καταστολή και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν γίνονται καθόλου σεβαστά στη χώρα αυτή. Παίρνουμε το στις 14 Αυγούστου ο Βασιλιάς είπε ότι θα ε, έθετε σε εφαρμογή κάποιες νέες διατάξεις, όμως τελικά τι έκανε μείωσε ακόμη περισσότερο τις ελευθερίες που υπήρχαν. Δεν ε, υπάρχουν ελευθερίες για τους πολίτες. και μάλιστα ε, τους στερούν και την πολιτική τους ταυτότητα στους πολίτες. Πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας για να υπάρχει ελευθερία του τύπου στη χώρα αυτή. Ας δούμε τι θα γίνει. Ελπίζουμε ότι στο Μπαχρέιν θα ληφθούν υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι πολύ σημαντικό για να προωθούν οι μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Γκέριγκερ Δεόντεμπεργκ. 1,5 λεπτό συνάδελφο Σάκε. Πρόεδρε και Επίτροπε, ακόμη μια φορά χρειάζεται να ασχοληθούμε με τον Μπαχρέιν. Πρέπει βέβαια να συγκρίνουμε και με την κατάσταση της Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία συμβουλεύει τον Μπαχρέν και του χορηγεί ακόμη και άρματα. Αντί όμως να ζητήσουμε διάλογο ή την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, βλέπουμε ότι ο βασιλεύς του Μπαχρέιν έχει απαγορεύσει κάθε διαδήλωση. Δεν είναι όλοι οι αντιφρονούντες τρομοκράτες ή πράκτορες του Ιράν. Και δεν πρέπει να επιτρέπεται ποντεβασανιστήρια υπό ιεσδήποτε συνθήκες. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει μία έρευνα για την κατάσταση στο Μπαχρέιν που πρέπει να απελευθερώσει αμέσως τους πολιτικούς κρατουμένους ιδίως όσους έχουν ενωσιακή υπηκότητα. Πρέπει και οι δύο πλευρές στο Μπαχρέιν να αρχίσουν διάλογο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να είναι ελεύθερα γιατί αυτή τη στιγμή είναι πολύ πολλωμένα και ο ειδικό συζητητής για τα βασανιστήρια δεν του έχει χορηγηθεί άδεια να ερευνήσει. Δυστυχώς επίσης με τη βοήθεια ενωσιακής τεχνολογίας χρησιμοποιούνται λογισμικά για να παρακολουθούν τους αντιφρονούντες οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν πρόκειται να βοηθήσουν και ελπίζω εμείς και ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο να εκφράσουμε στεναρότατα τη στάση μας για την καταδίκη της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Μπαχρέιν. Ευχαριστούμε κυρία Σάκε και τώρα για ένα λεπτό ο συνάδελφος Μπίλαν. Ευχαριστώ. Πρόκειται για μια ακόμη χώρα της Μέσης Ανατολής, ε, όπου είδαμε μια πολύ αιματηρή καταστολή των δημοκρατικών ε, διαμαρτυριών από την κυβέρνηση. Και βλέπουμε πως αυτό το ειδικό δικαστήριο το οποίο ουσιαστικά ασχολείται με την καταστολή των διαδηλωτών, ε, πώς λειτουργεί πρέπει να κάνουμε μια έκκληση στην κυβέρνηση του Μπαχρέιν για να σέβεται τους διαδηλωτές και να υπάρχει και ελευθερία του τύπου των μέσων ενημέρωσης. Επίσης ε, θα πρέπει να απελευθερωθούν ε, οι πολιτικοί κρατούμενοι και να υπάρχει και ένα δίκαιο δικαστικό σύστημα. Ο Υπουργό ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι καλό, ναι, αλλά πρέπει να συνεχίσει η άσκηση πίεση στο Μπαχρέιν. Πρέπει να υπάρχει πίεση από τη διεθνή κοινότητα για να γίνεται για να υλοποιούνται οι μεταρρυθμίσεις. Ελπίζω να μας ακούνε κάποιοι εκεί στο Μπαχρέιν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπίλερ. μισή λεπτό ο κύριος Μέρφυ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως και εκατομμύρια ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο, οι νέοι και οι εργάτες ε, στο Μπαχρέιν εμπνεύστηκαν από τις επαναστάσεις στην Τινησία και στην Αίγυπτο και θέλησαν να, ζητήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα, να ζητήσουν δημοκρατικές συνθήκες. Αλλά όταν ε, ζήτησαν αυτά τα δικαιώματα, συνάντησαν ε, την άγρια καταστολή των ε, ενόπλων δυνάμεων του Μπαχρέιν. Σχίζει αυτή η καταστολή ε, και έναντι ε, δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Πολλοί από τους δημοσίους υπαλλήλους έχουν προσαχθεί διότι ε, έλαβαν μέρος σε διαμαρτυρίες. Οι 31 από τους 48 εργαζομένους στον τομέα της υγείας ε, ε, δεν είχαν τη δυνατότητα να επανέλθουν στην θέση εργασία τους μετά τις διαμαρτυρίες. Τον Αύγουστο ο βασιλιάς Σαμάντ εξέδωσε ένα διάταγμα που περιορίζει την ελευθερία του συνέρχεστε στο κέντρο της πρωτεύουσα. Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν διότι απλώς ασκούσαν το δικαίωμά τους στην, στο να διαμαρτυρηθούν θα πρέπει να αποκατασταθούν ως προς τα δικαιώματά τους. Πρέπει να ρωτήσουμε πόσο υποκριτικό είναι αυτό το θέμα το ότι αυτοί οι οποίοι, οι δυνάμεις αυτές οι ε, οποίες ε, καταδικάζουν την κατάσταση στη Συρία, οι Ηνωμένε Πολιτείες και Γαλλία ε, έχουν εμπόριο όπλων με αυτή την περιοχή του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μέρφη και κύριο Όμπερ Όμπερμαγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και στο Μπαχρέιν η δημοκρατική άνοιξη ε, βρήκε υποστηρικτές. Δυστυχώς όμως στο Μπαχρέιν οι πολίτες ε, δεν είχαν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τα αιτήματα της 21ης χιλιετίας γιατί η βία και η καταπίεση και η καταστολή τους εμπόδισαν ε, το Μπαχρέιν είναι πολιτική και οικονομική εταίρη της Δύσης και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βλέπουμε ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, υπενθυμίζω μια δήλωση του Κόφι Ανάν ε, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έλεγε ότι οι παραβίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του σήμερα είναι οι σφαγές του αύριο. θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και αν δεν υπάρξει ε, κάποια συμμόρφωση θα πρέπει να υπάρξει και τιμωρία, εμπάργο και ε, διακοπή οικονομικής βοήθειας και συνεργασίας. Θα πρέπει λοιπόν σύμφωνα με αυτά τα οποία πρεσβεύουμε να πράττουμε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπερμάγκερ και τώρα συνεχίζουμε με τους ομιλητές, με την κυρία Κορόλα. Ευχαριστώ. Δεν ε, είναι εύκολο να ασκείται πολιτική υπό την ε, επιρροή των ΗΠΑ, της Σοβιτικής Αραβίας ε, και του Ιράν. Πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι και η κυβέρνηση του Μπαχρέιν είναι δύσκολο να καταπολεμήσει τις ταραχές ε, σε ένα τέτοιο πολιτικό περιβάλλον. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν ανησυχώ για την κατάσταση εκεί η κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει το δικαίωμα ε, της ε, συγκέντρωσης, της συνάθρησης, όμως ε, θα πρέπει να επιτρεπεί στους ανθρώπους να μπορούν να συνεθρίζονται. Εγώ ανησυχώ για το πώς αντιμετωπίστηκαν οι διαδηλωτές και επίσης ποια ήταν η μεταχείριση που επιφυλάχθηκε σε όσους προσέβαλαν τον βασιλιά. Ελπίζω όμως να μπορέσουμε να βρούμε ειρηνικέ λύσεις για την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βανόντεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Μπαχρέιν είναι φίλος και σύμμαχος. Έχει μια γεωστρατηγική σχέση κλειδί στον Περσικό κόλπο. Ε, είναι ε, κέντρο ε, δράσης για τον Πέμπτο Στόλο και είναι στενός σύμμαχος της Σαουδικής Αραβίας. Όλοι αυτοί είναι παράγοντες που κάνουν τον Μπαχρέιν στόχο αποσταθεροποίησης στην περιοχή και στόχο για όσους θέλουν να πλήξουν τις σχέσεις με, την, με τη Δύση. Σίτες και Σουνίτες ζούσαν ειρηνικά επί χρόνια. Τώρα βλέπουμε ότι είναι αντικείμενο εκμετάλλευση αυτέ οι διαφορέ. Και βεβαίω υποστηρίζουμε το δικαίωμα σε διαμαρτυρία και το δικαίωμα ε, του συνέρχεστε και οι πρωτοβουλίες του Βασιλιά όσον αφορά τον εθνικό διάλογο και τις ε, ε, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κινήσεις που πρέπει να χαιρετήσουμε αλλά παράλληλα πρέπει να δούμε και τις τρομοκρατικές πράξεις που έχουν διαπραχθεί και θα συνεχίσουν να υπάρξουν προκλήσεις ε, στους δρόμους του Μπαχρέιν και τα μέσα ενημέρωσης θα προσπαθούν να αναζητήσουν ε, ρεπορτάζ βιαιότητας ε, και βίας. Νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι είναι αντίθετοι με τις τωρινές πολιτικές ρυθμίσεις θα καταδικάζουν την τρομοκρατία και τη βία και θα συμμετάσχουν δημιουργικά στο διάλογο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βανόρντεν. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Συνάδελφος Κέλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ειλικρινά το Μπαχρέιν δεν είναι σε τόσο άσκημη κατάσταση όπως άλλες χώρες που συζητήσαμε εδώ μέσα και πρέπει να αναγνωρίσουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί εκεί ιδιαίτερα σε, άμα σκεφτούμε ότι δημιούργησε τη θέση του διαμεσολαβητή για την αστυνομία. Επίσης είναι κάτι που δεν γίνεται συχνά στις χώρες εκείνες. Αν υπάρχουν αδυναμίες αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να πιέσουμε τον Μπαχρέιν για την ελευθεροτυπία ιδίω που είναι σημαντικό στοιχείο για οποιαδήποτε χώρα για τη χρήση των κοινωνικών μέσων και γενικά για την πάυση των φυλακίσεων των αντιφρονούντων. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλη μου. κύριε Κρετού. Ευχαριστώ Πρόεδρε μετά τις δράσεις της κυβέρνησης της Μανάμα και μετά την διεκαταστολή των διαδηλώσεων Βλέπουμε ότι δεν τηρούνται τα δικαιώματα του συνέρχεσθε. Θα πρέπει να ζητήσουμε να μπει ένα τέλος ε, στις διώξεις και στις ε, καταχρήσεις. Ε, να επιτραπεί στους πολίτες να κινούνται ελεύθερα και να έχουν το δικαίωμα του συνέρχεσθε. Επίσης θα πρέπει να έχει πρόσβαση στη χώρα ο ειδικό εκπρόσωπος για τα βασανιστήρια και για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να αποκατασταθεί το σύστημα δικαιοσύνης στο Μπαχρέιν έχει επιλεγεί τον Μπαχρέιν ως έδρα του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αυτό είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, είναι μια πρωτοβουλία του Αραβικού Συνδέσμου και το χαιρετίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Κρέτου. Συνάδελφος Πάσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε συμφωνώ ότι όταν διατυπώνουμε τα αιτήματά μας προς τον Παχρέν θα πρέπει να είμαστε επικοδομητικοί. Θέλουμε να ζητήσουμε κάποιες αλλαγές, αλλά παράλληλα θα πρέπει να γνωρίζουμε και τα ε, μέρη στα οποία απευθυνόμαστε. Υπάρχουν Ισλαμιστές, υπάρχουν δημοκρατικές δυνάμεις. Στο Μπαχρέιν μπορεί να γίνει διάλογος με την κυβέρνηση και με τον βασιλιά. οι κινήσεις που έχουν γίνει, το ότι έχει οριστεί υπεύθυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μεσολαβητής δείχνει ότι υπάρχει κίνηση προς ε, την απελευθέρωση, ε, προς την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης ε, και προς τις ελευθερίες των πολιτών. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Εσαγιά. Ευχαριστώ. Η κατάσταση στον Μπαχραήν αποτελεί αποτέλεσμα του ξεσηκώσμου της Αραβικής Άνοιξης και η κυβέρνηση για να ελέγξει την κατάσταση προσπάθησε να περιορίσει τα θεμελιώδη δικαιώματα για τις πολιτικές ελευθερίες. Προκειμένου όμως να ελεγχθεί η τρομοκρατία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται υπερβολική βία και όσοι διαπράττουν ε, ε, αδικήματα θα πρέπει να οδηγούνται ενώπιος της δικαιοσύνης. Υπάρχουν βέβαια χώρες ε, σε αυτήν την περιοχή με χειρότερη κατάσταση, που βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση σε ό,τι αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι η χώρα αυτή έχει σημειώσει πρόοδο. Λυπούμε που δεν θέλουν όλες οι πολιτικές ομάδες να υποστηρίξουν αυτό το ισορροπημένο κείμενο. Ολοκληρώνεται η διαδικασία Catch the Eye και δίνουμε το λόγο στην Επίτροπο Πρόεδρε, Εξ αρχής θα τονίσω ότι η κατάσταση στο Παχρέιν ε, είναι ανησυχητική. Η Αντιπρόεδρος Άστον μου ζήτησε να κάνω ακριβώς αυτή τη δήλωση εδώ. Η Αντιπρόεδρος Άστον παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την κατάσταση ε, στον Παχρέιν από την αρχή των ε, ταραχών το Φεβρουάριο του 2013 και έχει έρθει σε επαφή με τις αρχές και με τον βασιλιά και με την κοινωνία των πολιτών στο Μπαχρέιν. Ακόμη θα ήθελα ε, να τονίσω ότι προς όλες τις πλευρές ε, τονίζουμε ότι πρέπει να σταματήσει η βία και να οδηγηθούν ε, στην εθνική συμφιλίωση. Αυτό πρέπει να είναι το βασικό μας μέλημα. Η Αντιπρόεδρος Άστον ζήτησε από τον Σταύρο Λαμπρινίδη, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, να κάνει μια επίσκεψη στο Μπαχρέιν πριν τη δική της επίσκεψη για το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου στις 13 Ιουνίου. Και στην επίσκεψη αυτή ο κ. Λαμπρινίδης συνάντησε εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, της κοινωνίας των πολιτών, επισκέφθηκε ε, φυλακισμένους που κρατούνται για πολιτική δραστηριότητα και επανέλαβε ότι η διαδικασία συμφιλίωσης απαιτεί και μετριοπάθεια και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης από όλες τις πλευρές θα πρέπει αυτό να συμπεριλαμβάνει την απελευθέρωση αυτών που συνελήφθησαν στο πλαίσιο ειρηνικών διαμαρτυριών και αυτό είναι προϋπόθεση για να μην υπάρξει πόλωση της κοινωνίας στο Μπαχρέιν. Η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν παραμένει σήμερα ένα σημαντικό θέμα και η διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης θα πρέπει να κάνει πολλά βήματα. Ζητούμε από τις αρχές να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι νόμοι θα είναι συμβατοί με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να προστατεύονται και να τηρούνται στην πράξη. Κατά τις τελευταίες μέρες εκφράσαμε τις ανησυχίες μας στους ομολόγους μας στο Μπαχρέιν σχετικά με νέα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην άρση της ε, ηθαγένειας ε, και στη ρύθμιση των επαφών μεταξύ ε, πολιτικών ομάδων και διπλωματικών αποστολών. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. Θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τον Μπαχρέιν να εφαρμόσει πλήρως ε, τις συστάσεις ε, της Επιτροπής Περιοδικού Ελέγχου και Παρακολούθησης. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αυτή την κατεύθυνση γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να οδηγήσει σε μια βιώσιμη διαδικασία μεταρρύθμισης. Ε, τον Ιούλιο χαιρετήσαμε το ότι υπάρξει ένας διαμεσολαβητής για την αστυνομία και θα συνεχίσουμε να τονίζουμε ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η ατιμορρησία. Αυτή η νέα μονάδα μαζί με την εισαγγελία θα πρέπει να εκπληρώσουν το καθήκον τους με πλήρη ανεξαρτησία. Εποφελούμε της ευκαιρίας για να χαιρετήσω την κοινή δήλωση για τον Μπαχρέιν όπως εκφράστηκε στο Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκεμβρίου και όπως υποστηρίχθηκε από όλα τα κράτη-μέλη. Χαιρετίζουμε και την συνεισφορά της αντιπροσωπείας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Αραβική ε, Χερσόνησο ε, τον Απρίλιο του 2013 κατά την επίσκεψη στο Μπαχρέιν και πιστεύω ότι είναι πολύ ισορροπημένο το ψήφισμα στο οποίο καταλήξατε. Ευχαριστούμε την Επίτροπο Ρέντινγκ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση λοιπόν. Έχουμε έξι προτάσεις ψηφίσματος και θα ακολουθήσει άμεσα η ψηφοφορία. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω. Έχουμε ένα διαδικαστικό θέμα.